Καλησπέρα. Δεν είμαστε υπεράριθμοι, αλλά είμαστε παρκείς. Η συνέλευση και στην ε, Κοπενχάγη μας αφαιρεί μέλη. Η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται μέσω του ίντερνετ. 16 Μαΐου έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Έχουν γίνει μερικές τροποποίησεις, τις έχουμε ανακοινώσει. Λείπει και η κυρία Γιατερμέκη, η οποία μας ζήτησε να εξετάσουμε ως αριθμό 1 το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, της οποία... του οποίου είναι η συγγήτρια. Αν φυσικά συμφωνείτε. Επίσης η έκθεσή μου που αφορά στα άρθρα 20, 27 και 50 θα αναβληθεί για μία επόμενη συνεδρίαση. Γιατί και το Προεδρείο θέλει να πει τη γνώμη του. Ήρθα σε επαφή και με τον Πρόεδρο, δεν υπάρχει τίποτα το επίγον, άρα περιμένουμε. Εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Και πάμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου. Το τμήμα θεματικών ερευνών μας έχει, στείλει ένα σημείωμα ενημερωτικό σχετικά για το καθεστώς επικύρωσης των ε, παρακάτω συνθήκων. <coughs> Συνθήκη για την ε, στραθερότητα, το Fiscal Compact, όπως επίσης και η συνθήκη που θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μας ενημέρωσε λοιπόν ε, η σχετική υπηρεσία ότι έχει τροποποιηθεί το άρθρο 136 για τη λειτουργία της, ε, για τη λειτουργία της Ένωσης. Τώρα έχουμε τα πρακτικά. Να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 20 12ου του 11, 19 23 του 12 και 17 Τετάρτου του 12. Έχετε τα πρακτικά στη διάθεσή σας και αν δεν έχετε παρατηρήσεις εγκρίνονται. Ήρθε στο μεταξύ η κυρία Γετερμέκη. Ήρθε, Ναι, σας είδα πρώτα και μετά σας ε, έχασα, διότι σας σκέπασε ο καφές, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, θελήσατε να εξετάσουμε ως πρώτο σημείο το σημείο 6, κώδικας διοικητικής διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να εξετάσουμε το σημείο. Ορίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου η κυρία Γιατερμέκη ως ε, εισηγήτρια και παρουσιάζει μία γνωμοδότηση. <coughs> σχετικά με έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Έχετε το λόγο κυρία Γιατερμέκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρώτη γιατί έχω και ένα άλλο θέμα σε άλλη επιτροπή. Θα μιλήσω όμως στην Φινλανδική. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για διαδικαστικές διαδικασίες, διοικητικές διαδικασίες για νομοθέτημα που βασίζεται δηλαδή στη συνθήκη της Λισαβόνας και συγκεκριμένα το, 200, το άρθρο 298 που απαιτεί από την Ένωση και τα θεσμικά της όργανα να εφαρμόζουν την λεγόμενη καλή διακυβέρνηση, χρηστή διακυβέρνηση. Το αναφέρει λοιπόν αυτό μεταξύ των αρχών η Ένωση. Είναι σημαντικό βέβαια θέμα όχι μόνο γιατί τέθηκε ενισχύ η συνθήκη αλλά και είναι σημαντικό και για τους πολίτες και τους υπαλλήλους της Ένωσης. Για τα όργανα και τους δημοσίους υπαλλήλους κυρίως, διότι το νομοθέτημα απαριθμεί ρητά ποιες είναι οι αρχές της καλής διακυβέρνησης στο παρελθόν δεν μπορούσαμε εύκολα να ταυτίσουμε παρατυπίες και παρανομίες. Είναι βέβαια σημαντικό και για τους πολίτες διότι μιλάει για τη διοντολογία της εργασίας των. Ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την νομιμότητα της ενωσιακής λειτουργίας και αυτό πολύ σημαντικό. Μπορεί μερικοί να διαβάσατε στην Herald Tribune τι λένε ορισμένα δημοψηφίσματα για την νομιμότητα της Ένωσης. Δυστυχώς δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ένωση. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν είναι βέβαια τίποτα το επαναστατικό και ξέρω ότι δεν έχουν τέτοιου είδου νόμους καλής διακυβέρνησης όλες οι χώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο το γνωρίζει ο Ανδρέας δίπλα μου, δεν υπάρχει τέτοιος νόμος σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας. Ε, υπάρχει όμως στις βόρειες χώρες και μάλιστα επισήμως. Δεν είναι όντω τίποτα το τελείως καινούριο. Στο, το, το 2001 ο διαμεσολαβητής ο ενωσιακός διαμεσολαβητής, συνέγραψε έναν κατάλογο αρχών δεοντολογίας που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Αλλά δεν ήταν βέβαια καμία δεσμευτική νομοθεσία. Υπάρχει και η χάρτα των θεμελιωδών που είναι δεσμευτική και που επίσης απαριθμεί ορισμένα δικαιώματα μεταξύ των οποίων την καλή ή χρηστή διακυβέρνηση και το δικαίωμα τα προβλήματα των πολιτών να μπορούν να επιλύονται νόμιμα και έγκαιρα. Πώς λοιπόν θα ανταποκριθούμε στα αιτήματα να είναι όλα αυτά τα όργανα ουδέτερα ανεξάρτητα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Αν έχετε όμως απορίες, με τα χαράς να σας τις λύσω. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ κυρία Γετερμέτικη. Ξεκινάει η συζήτηση. Ποιος θέλει το λόγο. Ο Ένιος ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν με λένε άνιου δεν καταλαβαίνω γιατί λέγομαι άγνιου λοιπόν. Α, άγνιου, α, άγνιου. Λοιπόν, η πρόταση αυτή για ελάχιστα πρότυπα που εκφράζεται εδώ ακούγεται σαν κάτι το πολύ επιτακτικό και είναι όντως περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερο κόστος για τους φορολογουμένους της Ευρώπης. Χρειάζονται βέβαια ποιοτικά πρότυπα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούν τα όργανα υποδειγματικά. Αλλά παρόλα αυτά, η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να βελτιώσει την εικόνα της Ευρώπης στα μάτια των φορολογουμένων, γιατί το βιωτικό τους επίπεδο έχει αμήλικτα μειωθεί από την Ένωση σε κάθε επίπεδο πολλά κράτη-μέλη διαπράττουν αυτή τη στιγμή ένα είδος αυτοκτονίας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση μπροστά ε, χωρών που ήταν κάποτε περήφανες. Κυρία Τάιν. Εγώ εκπλήσωμαι λίγο για τα όσα άκουσα μόλις από τον Βρετανό συναδελφό μας. Γενικά έχω κατανόηση για τις βρετανικές θέσεις που ζητούν μείωση του κόστους, αποδοτικότητα, αλλά στα πλαίσια της ε, διαδικασίας έχουμε ένα συνταγματικό πρόβλημα. Εγώ είμαι μέλος και στην Νομική Επιτροπή, όπου σε ομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο, που εργάστηκε και ήμουν και εγώ μέλος επί ένα έτος, εκεί οφείλω να πω ότι πραγματικά τρόμαξα που είδα ότι δεν έχουμε διοικητικό δίκαιο. Εκεί όπου διεξάγονται σημαντικές ε, δικαστικές διαδικασίες, έχουμε δηλαδή για τα καρτέλ για παράδειγμα, αλλιώς όμως τίποτα δεν είναι νομοθετημένο και για μένα αυτό είναι ακατανόητο. Αν έρθει ένας πελάτης, εγώ είμαι δικηγόρος και μου πει για μια διοικητική πράξη, για παράδειγμα, ότι θίγεται από μια διοικητική πράξη και δεν μπορώ να του πω εγώ ως δικηγόρος τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να αντιταχθεί, διότι δεν υπάρχουν νόμοι που να εξηγούν, που να λένε τι πρέπει να κάνει ο θυγόμενος. Γι' αυτό και προκαλείται μεγάλη σύγχυση και σε πολλούς τομείς δεν υπάρχει απολύτως καμία διαδικαστική διάταξη θεωρώ ότι αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Πώς θα διαμορφωθεί αυτό το δικονομικό δίκαιο και επειδή έχουμε 27 χώρες μέλη με πολύ διαφορετικές παραδόσεις στον τομέα αυτό, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει ο κατακαιρματισμός αυτός που οδηγεί, όπως είπα, να μην μπορεί κανεί να εξηγήσει τον πελάτη του περί τίνο πρόκειται, αλλά να υπάρξει ένα ενιαίο διαδικαστικό δίκαιο που να ισχύει για όλες τις διαδικασίες και για τους τομείς εκείνους όπου απαιτούνται ιδιαίτεροι κανόνες, όπως για παράδειγμα στο δίκαιο περί καρτέλ, ή για παράδειγμα πώς συμπεριλαμβάνεται ένα όνομα σε μια λίστα τρομοκρατίας ή πώς διαγράφεται, εκεί να προβλέπονται πρόσθετοι διαδικαστικοί κανόνες. Αλλά με τρόπο που να μπορώ να το εξηγήσω στον κάθε πολίτη και βεβαίως και τις προθεσμίες. Να γνωρίζει ότι για παράδειγμα μπορεί εφόσον θίγεται από μια πράξη της Κομισιόν να ε, προβάλλει ένσταση εντός ενός μηνός για παράδειγμα. Αυτό είναι πάρα οι πολίτες είναι απολύτως εκτεθειμένοι και δεν γνωρίζουν τι να κάνουν. Και αυτό βέβαια προκαλεί και τεράστια αλληλογραφία, διότι αν είμαι υποχρεωμένη να γράψω σε 10 διαφορετικές υπηρεσίες μέχρι να μάθω ποια είναι η πραγματικά αρμόδια, Όλα αυτά ε, προκαλούν μια έντονη δυσαρέσκεια. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα και νομίζω επίσης ότι υπάρχει ένα κενό κράτους, δικαίου. Υπάρχει ένα κενό εδώ στο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. κύριος Μπρόνς. Στην αρχή, ναι, Στην αρχή της έκθεσης παραδέχονται ειλικρινά ότι το κύριο πρόβλημα της Ένωσης είναι ότι οι πολίτες αμφισβητούν την νομιμότητά της. Ειλικρινές μεν, αλλά όχι αρκετά. Πολλοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλο και περισσότεροι, όντως αμφισβητούν την νομιμότητα της Ένωσης, μάλλον την αρνούνται, όχι απλώς την αμφισβητούν. Εκτός αυτού η νομιμότητα την αρνούνται, όχι γιατί δεν χορηγούνται οι υπηρεσίες με χαμόγελο ή γιατί δεν είναι υψηλής ποιότητας, αλλά οι αντιρρήσεις είναι πολύ βασικότερες. Ο κόσμος θέλει να του λένε την αλήθεια. Αν το έγγραφο α είναι το ίδιο με το έγγραφο β, τότε πρέπει να το δέχονται αυτό. Αν υπόσχονται δημοψήφισμα πρέπει να το κάνουν. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν ειρηνικά με τους γείτονές τους, όχι να υφίστανται τους νόμους που εφευρίσκουν οι γραφειοκράτες, δεν θέλουν να υφίστανται ούτε τους γειτονές τους. Αυτό είναι το πρόβλημα με την έκθεση κυρίας Γερισμάκη. Λέει ότι τα έγγραφα πρέπει να είναι ευνόητα, πολύ επαναστατικό για την Ένωση. Και έχει βέβαια απολύτως δίκιο. Ευχαριστώ. Daff. Ε, Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Η Αλεξάνδρα Τάιν μίλησε για βρετανικές θέσεις. Την διαβεβαιώ ωστόσο ότι τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται. δεν υπάρχουν βρετανικές θέσεις για το θέμα του διοικητικού δικαίου. Υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων από πλευρά των Βρετανών Ευρωβουλευτών για το θέμα αυτό. Προσωπικά θεώρησα την επίκριση του άρθρου 6 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επίκριση σε αυτό το άρθρο μια συμπληρωματική αρμοδιότητας που μιλεί για διοικητική συνεργασία ως ενδυνάμει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την εξασφάλιση ποιοτική νομοθεσίας και διακυβέρνηση. Νομίζω δε ότι οι συγγραφείς της συνθήκη της Λισαβόνα οφείλουν να επενεθούν για αυτό. Στην συνέλευση τότε είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το τι περιεχόμενο είχε η διάταξη αυτή. και ότι τελικά θα νομοθετούσαμε μέσω κανονισμών. Που νομίζω είναι και ορθή απόφαση, η οποία λήφθη μετά από μακρές συζητήσεις. Χαίρομαι λοιπόν που φαίνεται να κατευθυνόμεθα προς τα εμπρός στον τομέα αυτό. Εγώ νομίζω ότι προτιμώ να διαβάσω το σχέδιο στις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που δεν το έχω διαβάσει ακόμη, και ε, να δω πόσο προχωρεί. Και να δούμε σε αυτήν κάτι σχετικά ακριβώς με την έννοια της διοικητικής συνεργασίας όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλούμε μόνο για τους ε, θεσμούς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών διοικήσεων. σε ό,τι αφορά την διατύπωση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Έτσι νομίζω. Ας μην λησμονούμε επίσης ότι η πρόταση θα εξεταστεί προσεκτικά από τις Εθνικές Βουλές. Αφού θα είναι αφού θα έχουν την υποψία ότι ενδέχεται να καταπατήσει προνόμια τους και την αρχή της επικουρικότητας. Νομίζω λοιπόν να λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά να μιλήσουμε με την Κομισιόν να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν όταν πρόσφατα ήρθε να μας δει ο Επίτροπος Σεύκοβιτς το θέμα δεν τέθηκε τόσο ουσιαστικά. Εγώ πάντως θα ήθελα να πιέσω περισσότερο την Κομισιόν για να μάθω τι θεωρούν ότι είναι και αναγκαίο και εφικτό στον χώρο του Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου. Ευχαριστώ, Χέφνερ. Έχουμε συνηθίσει στην Επιτροπή εδώ να ανεχόμαστε διάφορες παρατηρήσεις. Αλλά επιτρέψτε μου κύριε Άγνιου και κύριε Μπρόνς να σας πω ότι πραγματικά δεν γνωρίζω εάν εξυπηρετείτε πράγματι τα συμφέροντα των πολιτών και φορολογουμένων σας όταν προσπαθείτε επί πέντε χρόνια να παίζετε τον ίδιο δίσκο εδώ στην Επιτροπή. Όποιο θέμα και να τεθεί εδώ, αμέσω βγαίνετε και λέτε Α, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειαζόμαστε νέε ρυθμίσει. Είμαστε αντίθετοι. Φοβούμαι ότι δεν έχετε καν κοιτάξει περί τίνο πρόκειται. Μιλούμε για νομική προστασία υπέρ των πολιτών. Μιλούμε για κλείσιμο κενών του δικαίου που πρέπει να κλειστούν για να είναι ξεκάθαρε οι διαδικασίε έτσι ώστε οι αρχές να είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Δεν πρόκειται για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων των πολιτών ή δημοκρατία. Πρόκειται για ένα αντικείμενο τελείω διαφορετικό από αυτά που συζητείτε εσεί εδώ. Και νομίζω ότι αξίζει, εν πάση περιπτώσει, τον κόπο και η παρούσα επιτροπή, αλλά και τα μέλη τη. Εσεί, βέβαια, εξαιρείστε, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στι συζητήσει εδώ. Αξίζει λοιπόν καλύτερη μοίρα. Ήμουν και εγώ μέλος στην ομάδα εργασίας για το EU Administrative Law, στην ομάδα εργασίας της Νομικής Επιτροπής, όπου εργαστήκαμε εντατικά πολλά απογεύματα. Συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση της κυρίας Γιάτεν Μάκη. Δεν έχω επί να πω τίποτα απολύτως, παρά μόνο να την υποστηρίξω. Θα συζητήσουμε βέβαια κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά πραγματικά αγανακτώ όταν ακούω τέτοιες αθεμελίωτες παρατηρήσεις που νομίζω ότι δεν προστατεύουν διόλου τα συμφέροντα των πολιτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της σοσιαλιστικής ομάδας συμφωνούμε με τους γενικούς ε, στόχους. Και ότι οι γενικοί στόχοι αυτής ε, της ε, πρότασης μας βρίσκουν σύμφωνους. Ποτέ δεν σταμάτησε να εντείνεται η διοικητική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μία επέκταση αρμοδιοτήτων με την αναθεώρηση των συνθήκων που ανέθεσαν άμεσα διοικητικές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράδειγμα ο ανταγωνισμός. Και πολλές νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Κομισιόν αρμοδιότητες οι οποίες ε, δεν εμπίπτουν στις εθνικές διοικήσεις. Αυτές οι αρμοδιότητες διευρύνθηκαν και με τη δημιουργία οργανισμών ε, σαν ε, αυτών για την εποπτεία για τα δημοσιονομικά. Έχουμε μια αχανή διοικητική εξουσία που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκεί διοικητικέ αρμοδιότητες και αναλαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις εναντί όλων των πολιτών που εντάσσονται στην, ε, ε, ε, στην νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολίτες την χάνουν των ιδίων δικαιωμάτων και των ιδίων υποχρεώσεων δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται από τους διοικητικούς κώδικες ε, των κρατών μελών. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και πιο αποφασιστικοί προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας ε, μία ενια διοικητική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τουλάχιστον να φτιάξουμε ένα πλαίσιο, μία αφετηρία για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτή τη διοικητική διαδικασία. Όχι για να μπερδέψουμε παραπάνω την ε, διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να της δώσουμε διαφάνεια, αντικειμενικότητα, προβλεψιμότητα, για να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες έναντι της, ε, που προκύπτουν μάλλον από τα διοικητικά μέτρα της Ένωσης και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο πιο φιλόδοξα σχέδια. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γέτερ Μέκη για να απαντήσει, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ένας διοικητικό κώδικας δεν είναι απλό πράγμα. Είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη δουλειά. Εσείς μας πληροφορήσατε για το κατά πόσο χρειάζεται ένας διοικητικός κώδικας και τις απαιτήσει τις οποίες εγώ συμμερίζομαι. Δεν θα ήταν χρήσιμο βέβαια να ξέρουμε εμείς τι θα περιέχει ακριβώς ο κώδικας, αλλά πρέπει τουλάχιστον να δούμε τι κάνει η νομική επιτροπή και αν υπάρχει συγχρονία στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, με εξέπληξαν οι Βρετανοί που είπαν ότι όλα αυτά καταλήγουν σε περισσότερη γραφειοκρατία και κόστος. Δεν το πιστεύω αυτό. Στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά σημαίνουν γραφειοκρατία και κόστος. Χρειάζονται ορισμένοι κανόνες δεοντολογίας. Καλό είναι. Έχω γύρω 8.000 όταν θέλουμε να γράψουμε τροπολογίες ας πούμε πως πρέπει να γίνονται και θα ήταν καλό και οι πολίτες να γνωρίζουν ποιες είναι οι διαδικασίες που ισχύουν στην Ένωση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτού του είδους τον διοικητικό νομοθέτημα. Όπως είπαν και άλλοι δεν πρόκειται για τίποτε το επαναστατικό, εγώ εξάλλου δεν είμαι επαναστάτρια. Θέλω απλώς να χορηγήσω μια νομική προστασία στους πολίτες και τους δημοσίους υπαλλήλους. Και γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε αυτές τις διατάξεις. Υπόθηκε ότι πρέπει οι προτάσεις να είναι πιο συγκεκριμένες. Ναι, μπορεί, αλλά αλλά δεν είχαμε να πούμε τίποτε παραπάνω από όσα σας εξέθεσα. Θα μπορούσα να είχα γράψει πολλές σελίδες. Γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για όλα τα σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολούμαστε ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Μπορούμε να τα πούμε πιο συγκεκριμένα, αλλά δεν πρέπει να τα αλλάξουμε τελείως. Αρκεί να είναι δεσμευτικά όμως και όχι απλώς δεοντολογία. Για το χρονοδιάγραμμα λοιπόν, η γραμματεία ξέρει καλύτερα ίσως. Άκουσα όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ότι η Νομική Επιτροπή ανέβαλε τη γνωμοδότησή της ή τις συνεδριάσεις της. Αυτά. Όχι, όχι και κάτι άλλο ακόμα προς τον αγαπητό μου φίλο Ανδρέα. Ξέρω ότι γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα τη συνθήκη της Λισαβόνας στο θέμα αυτό όμως θα ήθελα να πω ότι ισχύει αυτό που είπα, ότι δηλαδή στη συνθήκη της Λισαβόνας λέει μόνο χρηστή διοίκηση μέσα στην Ένωση. Δεν μιλάει για το πώς πρέπει να διοικείται το κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη έχουν δικούς τους κανόνες. Εδώ μιλάμε για τα δικά μας όργανα μόνο. Μάλιστα. Εγώ ρώτησα απλώς. Είπα ότι χρειάζεται πολύ λεπτομερής ανάλυση. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα λοιπόν, η νομική υπηρεσία ίσως να μπορέσει να μας δώσει το κείμενό της πριν τις 30 Ιουνίου ώστε να θέσουμε μια διορία κατάθεσης τροπολογιών μέσα στον Ιούλιο αλλιώς θα χρειαστεί αναβολή γενικότερα και για τις τροπολογίες και για την τελική ψηφοφορία. Ευχαριστούμε κυρία Γιατεμάκη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις έτσι θα κάνουμε. Λοιπόν θα περιμένουμε. Και πάμε τώρα στο σημείο 4 δηλαδή η τροποποίηση του άρθρου 181 του κανονισμού για τα πλήρη πρακτικά και του άρθρου 182 για την οπτικοακουστική εγγραφή των πρακτικών. Ενδιαφερθήκαμε γι' αυτό γιατί ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας ζήτησε να αλλάξουμε τον κανονισμό για οικονομικούς λόγους. Γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος στα πλήρη πρακτικά σε όλες, για να δημοσιεύονται τα πλήρη πρακτικά σε όλες τις γλώσσες και θα δούμε τι έχει να μας πει ο εισηγητής μας κύριος Χούτσεφ. Δεν ξέρω αν είπα καλά το όνομά σας. Καλά είπατε κύριε Πρόεδρε ότι θα ξαναμιλήσουμε για εξοικονομήσεις και οικονομικά, αλλά τώρα με κάπως διαφορετικό τρόπο. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο το Προεδρείο είχε αποφασίσει τα πλήρη πρακτικά να τηρούνται σε όλες τις γλώσσες. Και αυτό ήταν τμήμα μιας δέσμης μείωση του κόστους, να οργανθούν μάλλον αλλιώ τα πλήρη πρακτικά, για να γίνουν εξοικονομήσει και στην μετάφραση και στη διερμηνία. Εκτός αυτού, μετά από την έγκριση αυτή της δέσμης εξοικονομητικών μέτρων για τον πολιτισμό του 12, το Κοινοβούλιο ήδη άρχισε να μεταφράζει τα πλήρη πρακτικά μόνο στα αγγλικά. Θα αλλάξει λοιπόν σχετικά και ο κανονισμός εν καιρό το δέοντι. Η τροποποίηση του, κανονι... του άρθρου 181 δεν είναι κάτι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Έμαθα πώς έχει η κατάσταση μιλώντας με διάφορους επαΐοντες για το θέμα. Πώς έχει λοιπόν Το άρθρο 181 λέει ότι η μετάφραση των πλήρων πρακτικών σε όλες τις γλώσσες προβλέπεται. Συνήθως χρειάζονται 4 μήνες και 8,6 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό σε σύνολο 11. Από τότε που υπάρχουν μόνο στα αγγλικά τα πλήρη πρακτικά, σημειώθηκε και κάποιος κίνδυνος ε, υπονόμευσης της αρχής της πολυγλωσσίας. Επειδή όμως ήδη είχαμε εγκρίνει μέτρα εξοικονόμησης, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Τι προτείνω λοιπόν. Η μετάφραση σε μία μονογλώσσα θέτει σε κίνδυνο την αρχή της πολυγλωσσίας. Επειδή όμως είναι πολύ ακριβή η μετάφραση όλες τις γλώσσες, μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Προτείνω λοιπόν να υπάρχει ένα να υπάρχουν τα πρακτικά στις επίσημες γλώσσες, αλλά να μην μεταφράζονται αυτομάτως. Δηλαδή, να γίνει σεβαστή η αρχή της πολυγλωσσίας, απλώς και μόνο κρατώντας το πρωτότυπο κείμενο, χωρίς μεταφράσεις. Έτσι βέβαια θα μπορεί κανείς να μας πει ότι υπάρχει ένα είδος ε, εκλεκτισμού, αλλά τι να κάνουμε. Όσοι ζητούν ή θα ζητήσουν διορθώσεις του λόγου, των λόγων τους, πρέπει να το πράξουν ώστε να είναι πιστά τα πρωτότυπα πρακτικά. Και όποιος θέλει να ζητήσει μετάφραση έστω συνοπτική να μπορεί να το κάνει. Αυτός ο νέος τρόπος δημοσίευση των πλήρων πρακτικών θα επιφέρει μεγάλες εξοικονομήσεις, αλλά για να υπάρχει και διαφάνεια και να δίνεται η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, υπάρχει και η οπτικοακουστική εγγραφή με προφορική μετάφραση, διερμηνία δηλαδή σε όλες τις γλώσσες. Άρα πρέπει να αλλάξει και ο, το άρθρο 182. το οποίο προτείνω να λέει ότι ως εγγύηση για τη διατήρηση της αρχής της πολυγλωσσίας και της διαφάνειας οι εργασίες του Κοινοβουλίου θα εκπέμπονται σε πραγματικό χρόνο με διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Έτσι θα υπάρχει μια εγγραφή των εργασιών για όλους και σε όλες τις επίσημες γλώσσες και με τη χρήση ειδικευμένης τεχνολογίας θα υπάρχει πολυγλωσσικό web streaming ώστε να μπορεί κανείς να βρει τι υπόθηκε και πώς υπόθηκε και τη μετάφρασή του. και για σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτά θα εμφαίνονται και στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου για την τρέχουσα και την προηγούμενη συνόδου τουλάχιστον η εβδομάδα. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Προσπάθησα να αλλάξω το άρθρο 181 και το 182 έτσι ώστε να είναι τα πράγματα σαφή και καθαρά αλλά αν έχετε απορίες και άλλες προτάσεις να τις ακούσω. Ο κύριος Άγνιου. Thank you, thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλιστα, εγώ είμαι Βρετανός και μπορεί να πείτε ότι θα δεχόμουν να είναι όλα μόνο στα αγγλικά. Αλλά υπάρχουν 22 επίσημες γλώσσες και να υπάρχει μόνο σε μια γλώσσα, να υπάρχουν μόνο σε μια γλώσσα τα πλήρη πρακτικά, νομίζω ότι αυξάνουν το δημοκρατικό έλλειμμα που είναι γνωστό ότι υπάρχει στην Ευρώπη. Όσοι δεν μιλούν αγγλικά. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αν λοιπόν κανείς δεν μιλάει αγγλικά, ποια είναι η εναλλακτική λύση να πάει στο ίντερνετ για να μπορέσει να δει τι υπόθηκε εξ ονόματός του. Αλλά δεν είναι και όλοι στο ίντερνετ ή γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν όλοι πού να τα βρουν όλα αυτά στο ίντερνετ. Ποιος θα υποφέρει λοιπόν, οι πτωχότεροι, οι γυρεότεροι, οι περιθωριακότεροι και οι κουφοί βέβαια. Αν μόνο προφορικά υπάρχουν οι μεταφράσεις, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και στις φτωχότερες χώρες της Ένωσης θα υπάρχουν τα περισσότερα αρνητικά συμπεράσματα. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι η Ένωση δεν ενδιαφέρεται να μειώσει το δημοκρατικό της έλλειμμα. Βέβαια δεν το δέχονται καν πολλοί ότι υπάρχει, πάντως πρόκειται για υπαναχώρηση. Η βίβλος λέει για τον πύργο της Βαβέλ. ότι συγχύστηκαν οι γλώσσες και δεν μπορούσε ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλον. Ο κύριος Μπρόντς. Ο κύριος Ήλτσεφ αντιμετώπισε το δίλημα σεβασμού της πολυγλωσσίας ή εξοικονομήσεων. Κατάφερε δηλαδή να ζητήσει εξοικονομήσεις χωρίς όμως να θυσιάσει την αρχή της πολυγλωσσίας και γι' αυτό πρέπει να τον συγχαρούμε. Και δεν το λέω για αστείο. Εγώ ήμουν για πολλά χρόνια κάποιος που αναγνώριζε μόνο δύο γλώσσες, τα αγγλικά και τα ξένα. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να θεωρήσει ότι εγώ θα ήμουν υπέρ μιας μονογλωσσικής κατάστασης με τα αγγλικά. Ότι τα αγγλικά γίνονται lingua franca όλων των οργάνων. Αλλά δεν το δέχομαι αυτό. Θα ήθελα η γλώσσα μου να παραμείνει μία από τις εθνικές γλώσσες. Απλώς. Και όχι να γίνει διεθνής ένα είδος δηλαδή απλοποιημένων αγγλικών για διεθνή χρήση. Αν η Αγγλία κάποτε βγει από την Ένωση θα είναι βέβαια ακόμη πιο φοβερό να έχει αφήσει πίσω τη γλώσσα της. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντάφ. το 7 έπαιξα κάποιο ρόλο στη λήψη της απόφασης από την Ολομέλεια να απορριφθεί η πρόταση της ΑΦΚΟ τότε γιατί θεωρούσα ότι η διεύρυνση της Ένωσης χρειαζόταν κάποιο χρόνο ώστε οι νέες χώρες μέλη, ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο, να έχουν κάποιο περισσότερη δυνατότητα να βιώσουν την πολυγλωσία πριν καθορίσουμε ποια θα είναι η τελική μορφή η τελική τύχη των μεταφράσεων ή μη των πλήρων πρακτικών. Στη συνέχεια όμως άλλαξα γνώμη με βάση την εμπειρία μου και λόγω της ύπαρξης των νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την γρήγορη μετάφραση Συμφωνώ λοιπόν τώρα με την πρόταση του εισηγητή. Ως ιστορικό βέβαια δεν με βρίσκει σύμφωνο γιατί είναι μια ένδειξη παρακμής αλλά δυστυχώς νομίζω είναι απαραίτητο απαραίτητη η πλημελής αυτή λύση αλλιώς το Κοινοβούλιο θα έχει τεράστια προβλήματα. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντάφα η κυρία η Κωνστανς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ιτσερ που εξέτασε αυτό το τόσο λεπτό θέμα για τα τεχνικά και επίσημα θέματα ε, που αφορούν στην τροποποίηση του κανονισμού και που θίγουν ένα σημαντικό σημείο την πολυγλωσία της πολιτικής μας ένωσης το θέμα της γλωσσικής ποικιλότητα, το θέμα της ταυτότητας της Ένωσης. Αυτή η πρόκληση είναι ε, παρούσα στην έκθεση του συναδέλφου και υπάρχει και ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό για το Κοινοβούλιο είναι η αρχή της ε, υπευθυνότητας ε, που θα πρέπει να κρατήσουμε σε αυτήν την περίοδο κρίσης, όπου θα πρέπει να κάνουμε και οικονομίες και να περιορίσουμε τις δαπάνες μας, όποια και να είναι η φύση αυτών των απαντήσεων. Ε, βλέπω ότι πρόκειται περί στενοπού. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μια ισορροπημένη λύση σεβόμενη την πολυγλωσία και από την άλλη σεβόμενη την αρχή της ευθύνης και να είμαστε και ρεαλιστές. Η έκθεση λοιπόν έχει την τιμιότητα να προτείνει μια λειτουργική λύση. Ε, αξίζει τον κόπο να αναρωτηθούμε ειλικρινά γύρω από το θέμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ στην ΑΦΚΟ, αλλά και στις ε, ε, πολιτικές μας ομάδες για το θέμα της μετάφρασης του πρακτικού in extenso και να είμαστε και παιδαγωγικοί ε, στις πολιτικές μας ομάδες για να αποφύγουμε τα προηγούμενα επεισόδια. Πριν λοιπόν διατυπώσουμε μία τελεσίδικη απάντηση, Χρειαζόμαστε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να μην είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Υπάρχει μία πρόκληση ουσίας η οποία κρύβεται πίσω από αυτά τα τεχνικά ή επίσημα α, από αυτήν την τεχνική ή επίσημη βιτρίνα. Θα πρέπει λοιπόν να το, να το ε, παρουσιάσουμε στους συναδέλφους αυτό το θέμα της πολυγλωσσίας, ε, να το εξηγήσουμε και στους συμπολίτε μας, χωρίς όμως απ' την άλλη να, μην, να αγνοήσουμε τις προσπάθειες εξοικονόμησης ε, χρημάτων. Ευχαριστώ τον συνάδελφο που ήταν ακριβής. Θα ήθελα να έχουμε το χρόνο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε όλες τις επιπτώσεις Πολλοί συνάδελφοι εδώ στο Κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο υπερψήφισαν το θέμα της, της οικονομίας, ε, χωρίς όμως ε, να έχουν καθαρά στο κεφάλι τους ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στη μετάφραση, στη διερμηνία κλπ. <coughs> Θα ήθελα λοιπόν να εμπλουτίσουμε την όλη συζήτηση, να προχωρήσουμε, να εμπαθύνουμε στη συζήτηση, να συζητήσουμε και το θέμα της ανάγκης της πολυγλωσσίας αλλά και της δημοκρατικότητας στις συζητήσεις μας. Μέσερ Σμιτ. Tak formand. På det her specifikke tema, der tror jeg, jeg vælger at tale mit eget sprog, nemlig dansk. Øhm,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 έλεγα ότι είναι σημαντικό που μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα συνεχίσω όμως τα αγγλικά. Οι πολίτες της Ένωσης χάνουν το αίσθημα νομιμότητος της Ένωσης λόγω πολυγλωσσίας ή απολίας αυτής. Σίγουρα αν δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους τους εδώ για να μιλήσουν στη μητρική τους γλώσσα, το αυξάνει το αίσθημα αυτό της έλλειψης νομιμότητας. Η πρόταση αυτή θέλει να αντιμετωπίσει τον φόβο αυτόν, αλλά ξέρουμε όλοι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που είδαμε πριν, ότι όλοι όσοι μπορούν να μιλήσουν μία από τις μεγάλες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, θα το πράττουν και δεν θα, μιλούν, θα μιλάει κανείς άλλο στη μητρική του γλώσσα. Εγώ στην Ολομέλεια μιλάω πάντα τη μητρική μου γλώσσα για να φανεί και από τους εκλογείς το πώς δουλεύουμε. Ιδιαίτερα στην έκθεση Γκουαλτιέρη, Γκουαρνέρο μάλλον με συγχωρείτε, για τον προϋπολογισμό, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα περισσότερων ταπανών σε ορισμένους τομείς. Δεν είναι εδώ καλό να ζητάμε περικοπές για το θέμα αυτό της πολυγλωσσίας. Γιατί έτσι αυξάνεται το χάσμα μεταξύ εκλογέων και εκλελεγμένων. Η κυρία Τάιν. Ja, ich möchte meinen äh, Kollegen anschließen. Also ich bin Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους μου. Εγώ παρακολούθησα και μάλιστα διεύθυνα στις ε, διαδικασίες του τριμερούς διαλόγου στο Στρασβούργο για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πρόκειται βέβαια για εξαιρετικά ειδική γλώσσα. Εγώ βέβαια μπορώ να πω αυτά που θέλω σε μια γενική πολιτική συζήτηση στα αγγλικά. Αν όμως μπούμε σε λεπτομέρειες και βεβαίως αν είναι ακόμα περισσότερο σε νομική γλώσσα είναι πολύ δύσκολα. Ποιο από εμά μπορεί να εξηγήσει το εμπράγματο δίκαιο στα αγγλικά. Γίνονται λοιπόν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλωστε πολύ συχνά δεν είναι συγκρίσιμες καν οι ορολογίες. Δεν μπορεί κανείς να πει καν ότι μια μετάφραση είναι σωστή ή λάθος, διότι δεν υπάρχουν καν ειδικά ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με την ακριβή μετάφραση αυτών των κειμένων. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες δυνατότητες εξοικονόμησης ε, στο Κοινοβούλιο. Θα ήταν λάθος να γίνει η προσπάθεια να εξοικονομηθούν εκεί και ιδίως για τις οπτικοακουστικές διαβιβάσεις που είναι κάτι το οποίο οι πολίτες το παρακολουθούν σήμερα. Στην ψηφοφορία πράγματι στην Ολομέρεια δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα το τι ψηφίζουμε και γι' αυτό τάσομαι και εγώ υπέρ να έχουμε λίγο χρόνο, εάν αυτό είναι δυνατό, για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το πρόβλημα και να το μεταφέρουμε στις πολιτικές μας ομάδες και στις αντιπροσωπείες μας τις εθνικές δηλαδή. Ο Τάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από μια χώρα που έχει λιγότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπων μιλάνε τη γλώσσα τους και εδώ ποτέ δεν μπορώ να μιλήσω την γλώσσα μου στην Επιτροπή αυτή λόγω των παράξενων διαδικαστικών κανόνων που ε, ισχύουν εδώ. Δεν παραπονούμε όμω, διότι πιστεύω ότι έχοντα υπόψη και ενδεχομένε άλλε διευρύνσει στο μέλλον θα αυξάνουν διαρκώ οι γλώσσες και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι γιατί άραγε να δίνουμε το προνόμιο στον Μπρόνς να έχει τα αγγλικά ως κοινή γλώσσα. Ε, να παρηγορήσουμε λίγο και τους Γάλλους και Γερμανούς. Ας πούμε λοιπόν τρεις επίσημες γλώσσες, συν Ισπανικά και Πολωνικά, που είναι τουλάχιστον μία από τις Σλαβικές γλώσσες, και ο καθένας μετά θα πρέπει να κάνει την επιλογή του, να μάθει τουλάχιστον μία από αυτές τις γλώσσες. Και πάντα βέβαια θα μπορούμε να επικοινωνούμε με ε, ευγενικότητες να χάσουν το επίσημο καθεστώς τους. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε εξοικονομήσεις, εγώ θα προτείνω όλες όλα τα μέλη να έχουν ένα καταποκοπή ποσό με το οποίο να μπορούν να πληρώνουν τους βοηθούς τους και οι βοηθοί αυτοί να μεταφράζουν. Εννοώ τώρα βέβαια και στα καθημερινά το everyday business και όχι τις ε, ε, ακριβείς ε, βέρμπατη μεταφράσεις των παρεμβάσεων. Ο κύριος Σειρά μου τώρα να πω κάτι. Λίγα λόγια δηλαδή στη δική μου γλώσσα. Τη βουλγαρική που είναι αρκετά εξωτική βέβαια. Αλλά για να μπω και εγώ λίγο σε αυτή την πολυγλωσία. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι και εγώ ίδιος έχω δουλέψει σκληρά σε αυτό το σχέδιο έκθεσης και μάλιστα το υπέβαλα, το έθεσα λοιπόν στην ε, πρόσοχή σας μαζί με ένα ερωτηματολόγιο. Για τις οποίες ερωτήσεις βέβαια δεν έχω και οριστική απάντηση. Πιστεύω ότι, δεν πιστεύω καν ότι έχουν οριστική απάντηση αυτές οι ερωτήσεις. Και πρώτα, η χρήση διεθνών γλωσσών των χωρών μελών. Αυτό είναι βέβαια πολύ ευαίσθητο θέμα, το κατανοώ. Το κατανοώ απόλυτα. Δεύτερο, φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να διασυνδεθεί με ένα είδος απόλυτα ρεαλιστικής, λιτής ε, προσέγγισης που να μην έχει απολύτως κανένα συναισθηματισμό. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο, μια διέξοδο δηλαδή, και να λύσουμε το πρόβλημα. Όταν μιλούμε για την χρήση των γλωσσών, Βέβαια πάντα βλέπουμε μια δύσκολη κατάσταση. Για παράδειγμα, τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτοί είχαν μια ενιαία γλώσσα. Τώρα τις έχουν κάνει τέσσερις. Με τέσσερα ονόματα. Διότι οι Σέρβοι λένε, α, εμείς μιλάμε Σερβικά, οι Κροάτες Κροατικά, οι Βόσνοι Βοσνιακά, και ακόμα και το Μαυροβούνιο λέει τώρα ότι μιλάει μαυροβουνιακά. Είναι η ίδια, ωστόσο, γλώσσα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποκαλούνταν σερβοκροατικά. Τώρα, όταν θα έρθουν οι Κροάτες και άλλοι βουλευτές από τα Δυτικά Βαλκάνια, όλοι θα είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις για το γεγονό ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δική του γλώσσα. Ωστόσο, η έκθεσή μου δεν έχει ως πρόθεση να κάνει διάκριση είτε κατά είτε υπέρ οποιασδήποτε γλώσσας. Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν ότι θίγονται στο μέλλον. Αλλά, κοιτάξτε, θα εξοικονομήσουμε πολλά λεφτά. Επίσης πολύ χρόνο. Και ας μην λησμονούμε ότι πολύ λίγοι μιλάνε μόνο μία γλώσσα εδώ στον σύγχρονο κόσμο. Είπαν κάποιοι ότι τα φτωχότερα έθνη θα είναι σε μειονεκτική θέση. Αυτό δεν είναι αλήθεια όμως, διότι αυτοί όλοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Διότι εκεί πηγαίνουν ξένοι τουρίστες. Πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Εγώ στα 10 χρονών ήμουνα και μίλαγα ήδη ρωσικά. Και 18 είχα μάθει τα αγγλικά και 19 είχα μάθει κάποια γερμανικά και όταν πήγα στο στρατό, διότι εκεί είναι υποχρεωτική η στάτευση, χρειάστηκε να μάθω και τα τουρκικά. Να λοιπόν πώς εξελίχθηκε η ζωή μου. Και γνωρίζω από εμπειρία ότι είναι δυνατό να είναι κανείς πολύγλωσσος. Είπα προηγουμένως για εκλεκτισμό, στην αρχική μου δηλαδή παρέμβαση, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά αναπόφευκτο, διότι η παρεμβάσεις θα είναι πολύγλωσσες. Τα πλήρη πρακτικά δηλαδή των παρεμβάσεων θα είναι σε όλες τις γλώσσες. Θα απομαγνητοφωνούνται στην πρωτότυπη γλώσσα. Εάν κάποιος θέλει να τα διαβάσει στη γλώσσα τους, τότε μπορεί. Αυτά μπορούν να μεταφραστούν ένα χρόνο. Αναμένω λοιπόν βεβαίω τι έξυπνε και πρωτότυπε ιδέε που θα έχετε για να ε, βοηθήσετε να διαλευκάνουμε, να ε, ξεδιαλύνουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Ιλτσέφ. Το χρονοδιάγραμμα. Τώρα. Μέχρι 5 Ιουνίου τροπολογίες. ψηφοφορία 11-12 Ιουλίου. Α, όχι, όχι, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Έτσι, 5 Ιουλίου και μετά Σεπτεμβρίου. Νταφ. Η συζήτηση του σημερινού απογεύματο απεκάλυψε μια παρανόηση. επί της φύσεως των προτινόμενων μεταρρυθμίσεων. Η ιδέα δηλαδή ότι υπάρχει μια πρόταση που λέει δήθεν ότι η αγγλική γλώσσα θα πρέπει να προτιμηθεί είναι μια μεγάλη ανοησία. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Άρα, πριν να εξηγήσετε, να προσπαθήσετε να τα εξηγήσετε αυτά τα πράγματα στις πολιτικές ομάδες, διαβάστε πρώτα την έκθεση Ήλτσεφ και δεύτερο, λόγω της ευαισθησίας του γλωσσικού εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι είναι σκόπιμο να δοθεί περιθώριο στις ομάδες να εξετάσουν το θέμα. Και σε βάθος μάλιστα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτή η 5η Ιουνίου, 6 δηλαδή, που είπατε ως προθεσμία τροπολογία. Α, Ιουλίου, μάλιστα. Mm. Εντάξει τότε. Λάθος. Τότε κάνει ένα πρόβλημα. Αφού είναι 5 η ιουνιου 6 η δηλαδη που ειπατε ω προθεσμια τροπολογια α ιουλιου μαλιστα mm τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ούτω αποφασίζουμε. 5 Ιουλίου τα μεσάνυχτα για τις τροπολογίες. 11-12 Ιουλίου συζητάμε και 17 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε. Σημείο 5. Διαθεσμική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ε, για, τις, ε, για το χειρισμό των διαφαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Ο κύριος Χέφνερ έχει, είναι ο εισηγητής και έχει και το λόγο. Στα αγγλικά. Υπό το φως της συζητήσεως που μόλις έγινε, θα προσπαθήσω να τα πω στα αγγλικά, η ερμηνεία των όσων αποφασίζουμε είναι και θα είναι σημαντική και στο μέλλον. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό τα όσα έχουμε συζητήσει να είναι προσιτά στα πρόσωπα εκείνα που ίσως σε 20-30 χρόνια θα θέλουν να ε, εξετάσουν τι έγινε. Θα προσπαθήσω να τα πω στα αγγλικά, αν δεν καταφέρω θα τα πω στα γερμανικά. Άρα λοιπόν, μιλούμε για διαθεσμική συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την χρήση από πλευρά του Κοινοβουλίου και πρόσβαση εμπιστευτικών πληροφοριών που έχει στη διάθεση το Συμβούλιο. Είναι σαφές νομίζω σε όλες και όλους ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες και η διαφάνεια είναι πράγματα σημαντικά και θεμελιώδη για τη λειτουργία της δημοκρατίας και ενισχύονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι επίσης σημαντικό εμείς ως Ευρωβουλή, αν θέλουμε να κάνουμε χρήση των εξουσιών μας που θεμελιώνονται στην συνθήκη της Λισαβόνας και μας αναθέτουν το ρόλο του συνομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μαζί με το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή το Συμβούλιο και επίσης στα όσα συζητούνται σε διεθνείς διαπραγματεύσεις όπου συμμετέχει το Συμβούλιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ απαραίτητο. Ένας πολύ αναγκαίος όρος έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να κάνει τη δουλειά που του έχει ανατεθεί από τους πολίτες. Αυτή λοιπόν η διαθεσμική συμφωνία έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης από πλευράς διαπραγματευτικής ομάδας που την εντολή της έλαβε από τους Προέδρους Πολιτικών Ομάδων και τις οποίες ηγήθηκε ο κύριος Λένε. Προσωπικά δεν ε, πήρα μέρος σε αυτή τη διαπραγματευτική ομάδα, όπως προβλεπόταν αρχικά. Αυτό που μπορώ να κάνω λοιπόν σήμερα ή μάλλον αυτό που έκανα είναι ότι συνέταξα έκθεση για την έκβαση των διαπραγματεύσεων αυτών που ε, τις διεξήγαγε πραγματικά πολύ καλά ή εν λόγω διαπραγματευτική ομάδα για λογαριασμό της Ευρωβουλής. Δεν θα επαναλάβω τα όσα διαλαμβάνονται στην έκθεση. Νομίζω ότι είναι κατανοητά και σαφή. Όμως θα αναφέρω, ή μάλλον θα κάνω μια πολύ ε, απλή βασική εισαγωγή, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εξηγηθεί ότι ο τίτλος ίσως είναι παραπλανητικός, διότι ο τίτλος έχει ως εξή. Λέει δηλαδή ότι αναφέρεται σε έγγραφα που δεν υπάγονται στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αν αυτό ήταν απολύτως έτσι όπως λέει ο τίτλος δηλαδή, τότε θα υπήρχε ένα κενό ανάμεσα στα όσα ήδη έχουν μπει στη Διαθεσμική Συμφωνία του 2002 για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και σε άλλα έγγραφα που υποπίπτουν στην ίδια πολιτική αλλά εξωτερική πολιτική και όχι πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Έτσι λοιπόν, εμεί προβλέψαμε μια διάταξη στι διαπραγματεύσει, στην έκθεση αυτή βέβαια, ώστε για τι ενδεχόμενε εκείνες περιπτώσει όπου μπορεί να προκληθεί ένα κενό, η λύση να είναι μικτές συμφωνίες. Δηλαδή συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν κοινή πολιτική με συγχωρείτε, να τα ξαναπώ, λέει ο Μιλόν. Τα μπερδεύω λιγάκι αυτά, ε, τα γερμανικά με τα αγγλικά. Ξαναλέω λοιπόν, τα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίε πολιτική, κοινή εξωτερική ε, ασφάλεια και άμυνα, μάλλον εξωτερική πολιτική, αλλά όχι ασφάλεια και άμυνα, να υπάγονται σε αυτή τη συμφωνία. Και μόνο οι πληροφορίε οι οποίε αναφέρονται σε κοινή εξωτερική πολιτική ή μάλλον σε πολιτική ασφάλειας και άμυνας εκεί θα ε, επιβάλλεται η συμφωνία του 2002. Ταυτόχρονα αυτό που διαπραγματευτήκαμε η Ροδευτική Ομάδα είναι ότι θα επανεξεταστεί η Διαθεσμική Συμφωνία του 2002 και η διαπραγμάτευση αυτής της επανεξέτασης θα γίνει ήδη στη διάρκεια του 2012. Πέρα από αυτό τώρα, και αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα θέματα, δηλαδή να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογή αυτής της διαθεσμικής συμφωνίας. Τα άλλα βέβαια ήταν ομαλότερα ή τέλο πάντων εξευρέθη συνένεση ευκολότερα. Το Κοινοβούλιο νομίζω ότι κατάφερε πολλά. Μία διαφοροποίηση στην διαχείριση, αποθήκευση των εγγράφων, ε, σε σχέση με την διαβάθμισή τους, τις διάφορες διαδικασίες για την διαβάθμιση των προσώπων που έχουν πρόσβαση, security clearance, επίσης υπάρχει και ευθυγράμμιση με την Κομισιόν. Τα άκρος απόρριτα έγγραφα ε, δεν υπάρχονται στην ε, συμφωνία αυτή. Τώρα, έχουν πρόσβαση διάφοροι ε, εισηγητέ, συνεισηγητέ και οδησηγητέ και μέλη των επιτροπών αναλόγως της περιπτώσεως. Υπάρχουν και συμφωνίες για ασθενή συνεργασία που διασφαλίζουν ανάλογο επίπεδο προστασίας διαβαθμιών εγγράφων μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Αυτά δεν έχουν απολύτως ε, διευκρινιστεί ακόμα. Αλλά έχουν ξεκαθαριστεί μέσα στη Διαθεσμική Συμφωνία και το Κοινοβούλιο καλείται να προσαρμόσει τις διατάξεις του, τις εσωτερικές δηλαδή, σε αυτή τη συμφωνία. Δεν επιτύχαμε όλα όσα επιθυμούσαμε. Για παράδειγμα, δεν επιτύχαμε να υπάρξει επίσημη διαδικασία για την διευκρίνηση συγκρούσεων. Θα δούμε. Πάντως για ορισμένες προβλεπόμενες περιπτώσεις έχουμε βρει, έχουμε βρει λύσεις. Αυτά νομίζω χρειάζεται να εξηγηθούν σήμερα σχετικά με την έκθεση και τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στην ίδια την έκθεση και όπου πολύ ευχαρίστως θα ακούσω εγώ τώρα τις ερωτήσεις και σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την αξία των συναδέλφων. Ο κύριος Χάφνερ που είναι γερμανόφωνος μας μίλησε αγγλικά και σε πολύ καλά αγγλικά κύριε Χάφνερ τα κατάλαβα όλα. Τα αγγλικά σας είναι πολύ καλύτερα από πολλών συμπατριωτών μου. Σας συγχαίρω λοιπόν. Παρ' όλα αυτά Τώρα θα πείτε, τώρα βάζει την πλάκα ο Άγνιου πάλι. Όσο πιο συχνά παίζεται μια πλάκα, τόσο πιο πολύ μπορεί να γρατζουνιστεί. Λοιπόν, τι θα κάνει η Ένωση για τα εμπιστευτικά έγγραφα. Μπορεί μερικά από αυτά, γιατί πολύ λίγα είναι τα έγγραφα που είναι περιορισμένης διάδοσης μπορεί να πρέπει να τηρούνται μυστικά και άρα να υπάρχει μία εξαίρεση στην αρχή της διάδοσης, ελεύθερης διάδοσης πληροφοριών για το κοινό εφόσον η Κομισιόν, το Συμβούλιο και τα λοιπά έχουν δώσει σαφή λόγο για τον οποίο μπορεί να απαγορεύει τη διάδοση του γράφου. Γιατί δεν υπάρχει και ένας κανονισμός που να λέει ότι μετά από ορισμένο χρόνο, 20-30 χρόνια, απελευθερώνονται και αυτά τα απαγορευμένα έγγραφα όπως γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω είναι η γνωστή συνταγή της Ένωσης να μας κρατάει όλους μη ενήμερους για να μην είναι υπόλογοι και να κρύβουν από τους ε, φορολογούμενους τι συμβαίνει. Αυτό μου θυμίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΚΤΑ κρατιούνται μυστικά για πάρα πολλά χρόνια. Ενώ στη Βρετανία ανάλογα όργανα τηρούνται μυστικές συνεδριάσεις μόνο για 48 ώρες. Πολύ μεγάλη διαφορά. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε αυτό λοιπόν. Η έκθεση λέει ότι δεν θα απαιτείται ειδική άδεια για τη διάδοση εγγράφων που δεν είναι εμπιστευτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απαιτείται άδεια και για τα έγγραφα που ξεπερνούν αυτό το επίπεδο. εννοεί αυτό. Είναι δύσκολο βέβαια να γνωρίζουμε ακριβώς τις κατηγορίες, αλλά ποια θέματα μπορούν να θεωρηθούν εμπιστευτικά. Ποια είναι τα κριτήρια για να αποφασίσει κανείς ότι το α ή το β έγγραφο θα είναι εμπιστευτικό. Ποια είναι η διαδικασία που τα ορίζει όλα αυτά και ποια είναι τα κριτήρια για τη χορήγηση αυτής της κατηγοριοποίησης. Η έκθεση λέει ότι η πρόσβαση θα χορηγείται ανάλογα με το θέμα είτε για τους συντάκτες και τους κοιόδης είτε για τα μέλη των επιτροπών. Ερωτώ λοιπόν και πάλι τι είδους θέματα θα περιορίζονται μόνο στη γνώση των συντακτών και όχι των συναδέλφων. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ. Τι είδους. Μου φαίνεται ότι δεν ζητάει κανένας άλλο το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Χέφναρ να απαντήσει. Ακούστε αγαπητοί. Αυτά που λέτε εσείς Freedom of Information Act δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο, δεν θα έχουμε ακριβώς το ίδιο στην Ευρώπη. Αλλά η βασική αρχή της πρόσβασης της πληροφορία ισχύει σε κάθε περίπτωση. Μιλούμε για έγγραφα εδώ, τα οποία είναι εσωτερικά έγγραφα και έχουν διαφορετικές διαβαθμίσεις και νομίζω θα ήταν σωστότερο το ίδιο το Συμβούλιο να εξηγήσει τα περί των διαβαθμίσεων. Το Συμβούλιο βέβαια οφείλει να ακολουθεί τους γενικούς κανόνες που ισχύουν και εμείς ακολουθούμε την διαβάθμιση που δίνει το Συμβούλιο στα έγγραφα. Εάν δεν έχουμε λόγους να προσβάλλουμε τις αποφάσεις αυτές. Αυτό θα πω απαντώντας ε, γενικά στην ερώτησή σας. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο. Και ε, αλήθεια, ε, ε ο πρόεδρος, θα μπορούσαμε να ορίσουμε το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες 13 Ιουνίου. και να ψηφίσουμε 12 Ιουλίου. Εντάξει, Χέφνερ. Οπότε, τώρα, πάμε στο σημείο 7. 18η έκθεση, βελτίωση της νομοθεσίας, εφαρμογή των αρχών επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Η κυρία Ρέγνερ είναι η η συγγήτρια, δεν το είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, αλλά μέχρι τις 31 του μηνός είναι η κατάθεση των τροπολογιών. Θα ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια. Κυρία Ρέγνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή για πρώτη φορά επαρκή αριθμό χωρών που έχουν υποβάλει ένσταση για λόγους επικουρικότητας και ζητούν από τα Εθνικά Κοινοβούλια να παρέμβουν. Αυτό βέβαια ας μην μας παραπλανά. Η κατάσταση μέχρι τώρα βέβαια εμφανίζεται τελείως διαφορετική. Δηλαδή, όταν εξετάζουμε πόσα νομοθετικά σχέδια έχουν υποβληθεί μόνο 34 έχουν λάβει αυτήν την μομφή της επικουρικότητας, την ένσταση μάλλον της επικουρικότητας. Υπάρχουν βέβαια περισσότερες γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Βουλών, 211. Αυτό όμως σημαίνει ότι 211 οι 34 είναι σχετικά περιορισμένος αριθμός, δηλαδή οι Εθνικές Βουλές είναι αρκετά ικανοποιημένες με την διαδικασία και δεν προβάλλουν τόσο πολλές ενστάσεις σχετικά με την επικουρικότητα. Αυτό σημαίνει ή υπάρχει άλλος λόγος ότι δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια είναι τόσο φορτωμένα με το εθνικό έργο που δεν έχουν πράγματι επιληφθεί ε, υποθέσεις Και αρχίζουν τώρα να ασχολούνται περισσότερο και θέτουν των δάχτυλων επί των τύπων των ύλων. Θεωρώ ότι η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικότερα ποιοι είναι οι λόγοι. Γιατί δηλαδή είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός των ενστάσεων για την επικουρικότητα. Έχουμε αρκετά νομικά εργαλεία στη διάθεσή μας. Άρα, πρόκειται για αρκετά ρεαλιστική προσέγγιση να υπάρξουν δηλαδή guidelines, κατευθυντήρες γραμμές για τα εθνικά κοινοβούλια, για τους θεσμούς, έτσι ώστε να εξετάζεται η τήρηση της αρχής της και της αναλογικότητας. Αυτά χρειάζεται να τα υπομνήσουμε. Πάντως εγώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στα επιχειρήματα εκείνα τα οποία βλέπω να περιλαμβάνονται συχνά σε ενστάσεις επικουρικότητας. Ότι είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να εξεταστεί ποιο είναι ο λόγος ύπαρξης της ε, ένστασης επικουρικότητας. Δηλαδή, όταν γίνεται προσεκτικότερη ανάλυση του θέματος, διαπιστώνεται καμιά φορά ότι κρύβονται και λόγοι σκοπιμότητας. Όταν δηλαδή μια Εθνική Βουλή δηλώνει ότι δεν ικανοποιείται από μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξετάζονται η σκοπή. Και αυτό το θέτω εγώ στη γνωμοδότησή μου. Με ενδιαφέρει πολύ βέβαια να ακούσω τώρα τα σχόλιά σας. Ο Ο Πάολο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Ρέγνερ. για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και για όσα μας προτείνει. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. διότι αφορά στην αξιολόγηση την ίδια που κάνουμε εμείς στην επικουρικότητα, δηλαδή την αρχή καταμερισμού των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω γενικές παρατηρήσεις και ειδικέ παρατηρήσεις για το θέμα, για την έκθεση, ειδική παρατήρηση. Δεν θα πρέπει εμείς να επικαλούμεθα το πρωτόκολλο 30 της ε, συνθήκης του Μάστριχ, αλλά το 2 της Λισαβόνας που αφορά στην συνθήκη, στην συνθήκη η οποία ισχύει σήμερα. και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε την ουσία του θέματος. Πρέπει να βρούμε τα συγκεκριμένα υλικά κριτήρια τα οποία δικαιολογούν την παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Είναι διαδικαστικά κριτήρια, πρέπει να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια. Θα αναφερόμουν κατά συνέπεια στο πρωτόκολλο 2 και της λειτουργίας της Ένωσης και όχι στο 30 της συνθήκης του Άμστερνταμ. Αυτή η συνθήκη δεν αφορά μόνο σε αυτή τη γενική παρουσίαση της συναδέλφου Ρέγνερ. Υπάρχει και μια άλλη σημαντική πλευρά. Πώς να συνδεθούμε με αυτά τα εθνικά κοινοβούλια τα οποία τρέφουν ένα σχετικό πατερναλισμό. έναντι ημών. Δηλαδή, αν τα εθνικά κοινοβούλια δεν θέλουν να δίνουν προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά δικά μας θέματα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε εμείς ξαφνικά να πάμε και να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν. Είναι κυρίαρχα όργανα και πρέπει να αποφασίσουν πώς θα, κινηθούν, θα κινήσουν τις διαδικασίες τους. Τα εθνικά θέματα συζητούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να, να δώσουν την πρωτοκαθεδρία στα δικά μας ευρωπαϊκά όποτε θέλουμε εμείς. Και θα έπρεπε να αρκούν οι επιχειρηματολογίες του Συμβουλίου και της Κομισιόν, διότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να μας πούνε δεν μας δώσατε επαρκείς πληροφορίες, αναλυτικές πληροφορίες. και έλεγα μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να μας πούνε εμάς αυτό το πράγμα αλλά και εμείς μπορούμε να πούμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια δεν δίνουν προτεραιότητα ή δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι δικό τους. Πρέπει εμείς λοιπόν να συγκεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας και πρέπει να το υπογραμμίσουμε στην έκθεση στο γεγονός ότι η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να, να δίνει πλήρη αναφορά και αναλυτικές εξηγήσει στα Εθνικά κοινοβούλιο, Κοινοβούλια. Επαναλαμβάνω, η μορφή με την οποία το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο, ο τρόπος με τον οποίο το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο εξετάζει τα ευρωπαϊκά ζητήματα, είναι αρμοδιότητα του κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσουμε εμείς για τα δικά τους ε, προβλήματα. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο θα πρέπει να, να φροντίσουμε να δίνουμε επαρκείς και αναλυτικές πληροφορίες στα εθνικά κοινοβούλια και αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήματος. Τώρα, η άλλη πλευρά του ζητήματος που αφορά σε ένα θέμα ε, αρχή, ένα πιο φιλοσοφικό ζήτημα είναι το πώς θα ερμηνεύσουμε εμεί την αρχή της επικουρικότητας. Εγώ συμφωνώ και λέγω ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν αρκεί μόνο για να αυξήσει τις αρμοδιότητες των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Εθνικών Αρχών. Όχι, χρειάζεται επίσης και για να αυξήσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η αρχή της επικουρικότητας είναι μια ουδέτερη αρχή. Δεν λέει ότι έχει παραπάνω αρμοδιότητες η Εθνική, ε, ότι υπερέχει η εθνική αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής. Εμείς θα πρέπει να ορίσουμε την αρχή της επικουρικότητας ως ένα optimum, ως μια optimum αρχή, ουδέτερη. Αυτή είναι η αρχή της επικουρικότητας διότι δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή ή στην Εθνική Αρχή. Είναι μία ουδέτερη αρχή. Και το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι το καταλληλότερο για το optimum κριτήριο για την ανάλυση και την εξέταση ορισμένων ζητημάτων. Πρόκειται λοιπόν για μια ουδέτερη αρχή. Και μπορεί να, να, εμπλέκει είτε την διεύρυνση είτε τον περιορισμό των, των ευρωπαϊκών Ερμοδιοτήτων. Διότι η αρχή της επικουρικότητας είναι μία αρχή ουδέτερη από, πολιτικ... από νομικής πλευράς. Από πολιτικής πλευράς όμως χρησιμοποίησαν την αρχή της επικουρικότητας τα κράτη για να μειώσουν, να περιορίσουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγα λοιπόν ότι η αρχή της επικουρικότητας νόμι... είναι νομικά ουδέτερη, αλλά πολιτικά αποτελεί το μπαϊράκι των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ομοσπονδία. Έχει όμως ομοσπονδιακή διάσταση σε ορισμένα ζητήματα και σε κάθε ομοσπονδία <coughs> υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων και περιφερειακών όμως ε, αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν ε, λοιπόν διαλεκτικές συγκρούσεις μεταξύ εθνικών <coughs> και ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων. Έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο, είναι μια ουδέτερη αρχή και περιορίζει και διευρύνει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Είμαι πεπισμένος ότι η συνάδελφος Ρέγνερ σίγουρα θα αναφερθεί σε όλα αυτά. Τελευταίο σημείο και ολοκληρώνω. <clears throat> Δεν κατάλαβα πολύ καλά και ρωτώ την εισηγήτρια. Δεν καταλαβαίνω αυτή την ιδέα του να γίνεται μία σύγκριση μεταξύ επιπτώσεων και αρχή επικουρικότητας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η αξιολόγηση επιπτώσεων είναι ένα μέσο, δεν είναι μία αρχή. Είναι σαφές ότι η εκτίμηση επιπτώσεων είναι πιο ευρεία από την αρχή της επικουρικότητας, διότι λαμβάνει υπόψη άλλα στοιχεία. Από ότι δηλαδή η αρχή της επικουρικότητας. Ας πούμε οι επιπτώσεις ε, λαμβάνουν υπόψη άλλα στοιχεία. Δεν πρέπει να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των δύο. Πρέπει πάντα λοιπόν εμείς να επιστήνουμε την προσοχή ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κεντρικό ρόλο τον οποίο παίζει η αρχή της επικουρικότητας. Υποστηρίζω ότι υπάρχει τεράστια σύγχυση. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των επιχειρημάτων υπέρ της αρχής της επικουρικότητας και υπέρ εκείνων της αναλογικότητας. Υπάρχει μία διαφορά. η οποία δεν διαφαίνεται απόλυτα πάντα, μεν, αλλά διαφαίνεται σαφέστατα από τα κείμενα. Όταν μιλάμε για επικουρικότητα, μιλάμε για επίπεδα αρμοδιοτήτων. Και εμείς θα πρέπει να συζητάμε αν πρόκειται για αρμοδιότητα εθνική ή ευρωπαϊκή. Όταν μιλάμε όμως για αναλογικότητα, τι κάνουμε, εξετάζουμε αν τα μέσα τα οποία διαθέτουμε σε ένα από αυτά τα δύο επίπεδα είναι τα κατάλληλα ή όχι. Είναι λοιπόν διαφορετικά αυτά τα θέματα μεταξύ τους. Σίγουρα διαπλέκονται διότι άμα έχουμε δυσαναλογία μέσων Σίγουρα υπάρχει παραβίαση της επικουρικότητας. Αλλά η επικουρικότητα απαντάει σε ένα πρώτο ερώτημα. Ποιο είναι το επίπεδο. Η αναλογικότητα ξεκαθαρίζει την καταλληλότητα των μέσων που διαθέτουμε. Διαφέρουν λοιπόν τα δύο πράγματα μεταξύ τους. Η επικουρικότητα και η αναλογικότητα. Οπότε. Ξαναλέω, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Σίγουρα εμείς δεν παίζουμε τον πρώτο ρόλο, διότι δεν είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας. Αλλά θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην αρχή, επί της αρχής επικουρικότητας και κατά αυτόν τον τρόπο και αξία δίνουμε στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά δεν γινόμαστε και οι υπόγειοι προασπιστές των εθνικών κοινοβουλίων που ξέρουν να προστατεύουν τον εαυτό τους μια χαρά. Όσοι ήταν εθνικοί βουλευτές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ωραία που υπερασπίζονται τον αυτό τους στα εθνικά κοινοβούλια. Δεν χρειάζονται το δικό μας πατερναλιστικό καπέλο. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι σύμφωνοι να εξετάσουμε και πάλι το θέμα της επικουρικότητας, το θέμα των υλικών κριτηρίων που έθεσε η συγγήτρια, όπως και τα μέσα τα οποία διατίθενται εμείς ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιο συγκεκριμένα η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ήδη βγήκε και η πρώτη κίτρινη κάρτα. Τα εθνικά κοινοβούλια λοιπόν πρέπει να αρχίσουν να συνηθίζουν να έχουν μία κουλτούρα για ευρωπαϊκά θέματα. Δεν θα ήμουν καθόλου μα καθόλου απεσιόδοξος. Εγώ θα επανεπικέντρωνα το ζήτημα θα εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία αυτής της έκθεσης για να εκλεπτύνω την όλη έννοια της επικουρικότητας και να την ξεκαθαρίσω. Και για να καταστήσω κατανοητό ότι δεν πρόκειται περί συγχύσεως, ότι δεν πρόκειται για έναν πύργο της Βαβέλ που αναφέρουν οι συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο, κύριος Άγνιο εδώ θα είμαι πιο σύντομος πρόεδρε. Η λέξη επικουρικότης φαίνεται ότι είναι αγγλική, αλλά εγώ δεν την άκουσα ποτέ μέχρι τη συνθήκη της Μαστρίχτης. Αν πάει κανείς σε ένα βρετανικό χωριό διαλέξει 10 τυχαίους και πει τι είναι επικουρικότης, οι εννέα δεν θα ξέρουν καν τι σημαίνει και ο δέκατος θα νομίζει ότι πρόκειται για κάτι άλλο. Να πάτε σε σχολείο, να μαζέψετε τους δασκάλους και να τους πείτε τι είναι επικουρικό της, πολλοί θα κοκκινήσουν γιατί δεν θα ξέρουν τι σημαίνει. Τι σημαίνει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κάνει τη χάρη να αφήσει στις εθνικές κυβερνήσεις ορισμένες δικαιοδοσίες οι οποίες όμως θα έπρεπε να είχαν δοθεί από τις εκλογές και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εκπληκτικό ότι τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις τους παραπονούνται. Αν και οι περισσότερες από αυτές δέχονται τη συνωμοσία για να μην έχουν ευθύνη. Άμα δείτε ιστορικά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, κάποτε υπήρχαν 90 με 100 νομοθετήματα το χρόνο. Τώρα έχουν μειωθεί σε 20 με 25. Σε αυτόν το βαθμό η επικουρικότητα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Είναι απλώς ένας όρος που χρησιμοποιείται εδώ μέσα για να λέει στον κόσμο ότι όλα, είναι, όλα πάνε καλά και έχουν εξουσία, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν συμβαίνει καθόλου αυτό. Κύριε Τέιν. Πρώτα, επιθυμώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της και ιδίως για το ότι στην παράγραφο 4 θέτει όντω τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, δηλαδή γιατί έχουν εκδοθεί τόσο λίγες επιτυχείς γνωμοδοτήσεις, ενώ πέρασαν τρία χρόνια μέχρι ότου λάβουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα και ότι μια σχετική ανάλυση θα ήταν επιθυμητή. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι ανάλυση από την Κομισιόν μάλλον δεν θα αποδώσει αντικειμενικό αποτέλεσμα, διότι η Κομισιόν θα έχει σαφώ την τάση να τα άρει όλα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε ανάλυση, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή να ανατεθεί σε εξωτερικού φορεί ή να την κάνουμε και εμεί οι ίδιοι. Εμεί σκεφτήκαμε στην Νομική Επιτροπή να ε, ιδρύσουμε ειδικό τμήμα που να εξετάζει τα λεγόμενα follow-up των νομοθετημάτων. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι θα ήταν σωστό τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια να αναλυθεί από την Κομισιόν. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ, είμαι φανατική οπαδός της αρχής της επικουρικότητας και έχω μελετήσει κιόλα και πώς κινείται, πώς λειτουργεί στην δική μου χώρα, τη Γερμανία. Βέβαια, είναι ομοσπονδιακή χώρα και εκεί έχει ένα μειονέκτημα απέναντι σε άλλες συγκεντρωτικές χώρες, διότι εκεί στην δική μου περίπτωση δεν έχουμε μία ενιαία βουλή, αλλά πρώτα 16 διαφορετικές βουλές των ομόσπονδων κρατηδίων. Κάτι το οποίο οδηγεί σε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις. Επομένως η προθεσμία των 8 εβδομάδων είναι στην ουσία πάρα πολύ περιορισμένη. Ασχολήθηκα και στο πανεπιστημιακό επίπεδο με τις ε, ιστορίες αυτές. Στη Γερμανία μπορώ να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Χρειάστηκε να περάσει πολλή χρόνος μέχρι ότου να αντιληφθούν και οι χώρες μέλη ποιο διαβιβάζει ποιο έγγραφο σε ποιον, ποιο λαμβάνει ποιο κτλ. Και μέχρι ότου αυτά περάσουν στην νομοθεσία. Ανεξαρτήτω μάλιστα από, τις, ε, από το μέγεθος των ομόσπονδων κρατηδίων εγώ είμαι από το Βερολίνο και είναι μικρή είναι μικρό ομοσπονδιακό κρατήδιο, Ομόσπονδιακό κρατήδιο μάλλον. Οπότε χρειάστηκε πάρα πολύ ε, καιρό, χρειάστηκε εννέα μήνες μέχρι ε, να κάνουμε αυτό το ξεδιάλειμμα. Διαπιστώσαμε εν τέλει ότι δεν λειτουργεί καλά αυτή η υπόθεση της επικουρικότητας. Εγώ με υπέρ του συστήματος APEX. Δεν ξέρω βέβαια αν τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα όλοι εδώ στην αίθουσα, διότι ακριβώς επειδή έχουμε διαπιστώσει Κάποιο πριν είπε ότι οι πόροι δεν είναι σπουδαία υπόθεση, αλλά οι μικρέ χώρε δεν έχουν του πόρου και ούτε καν πληροφορούνται τι γίνεται εδώ στι Βρυξέλλε. Πολύ λιγότερο μάλιστα να μπορούν να κάνουν και τι σχετικέ γνωμοδοτήσει. Έχουμε λοιπόν μια ιστοσελίδα εδώ και ένα εξάμεινο όπου δημοσιεύουμε τις γνωμοδοτήσεις αυτές και έτσι επιτρέπουμε στις μικρές χώρες μέλη να δουν «Α, μια στιγμή εδώ μια μεγάλη χώρα μέλος όπως η Γερμανία, όπως η Μεγάλη Βρετανία που η Μεγάλη Βρετανία κάνει πάρα πολλές ε, ε, ενστάσεις για την ειδικορικότητα, Έτσι λοιπόν οι χώρε μέλη δεν χρειάζεται οι μικρέ να κάνουν τον κόπο να τι γράψουν μόνε του τι ενστάσει αυτέ, αλλά μπορούν να πούν, α συνυπογράφουμε αυτή της ε, μεγάλη Βρετανία και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν να αφιερώσουν ειδικού πόρου. Αυτή πάντω η σελίδα Apex είναι λίγο πολύ άγνωστη. Εγώ με κάθε ευκαιρία την προπαγανδίζω και σε άλλες πολλές χώρες είναι άγνωστοι. Θα ήθελα να ρωτήσω και το Συμβούλιο, ρώτησα μάλλον στο Συμβούλιο και εκεί πολλοί δεν τα γνωρίζουν. Είναι λοιπόν καθήκον δικών μας των Ευρωβουλευτών να επισημάνουμε την ύπαρξη αυτής της ιστοσελίδας που θα επιτρέψει σε μικρές και μεσές ε, χώρες μέλη να μπορέσουν να συνυπογράψουν ενστάσεις μεγάλων χωρών. Εγώ πιστεύω προσωπικά, τουλάχιστον μπορώ να το αποκλείσω για την γερμανική Bundestag, ότι νομοθετήματα τα οποία δεν επιθυμούμε να δούμε για οποιουσδήποτε ουσιαστικού ή λόγου σκοπιμότητας να προσπαθήσουμε να τα πετάξουμε έξω επικαλούμενη την ε, επικορικότητα. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνω. Βέβαια, εμείς βρισκόμαστε πάντα στα όρια της νομιμότητας. Δεν έχω αντίρρηση για την αρχή της επικουρικότητας. Εξετάζω κιόλας για τους νόμους για ποιο λόγο είναι αρμόδιο το ευρωπαϊκό επίπεδο και για ποια πράγματα είναι αρμόδια τα εθνικά επίπεδα. Εκεί βέβαια για την διάκριση αυτή, για παράδειγμα ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκαιο αγοραπολισιών, είναι υπόθεση της ε, νομικής μας επιτροπής. Αυτά δεν ε, βασίζονται άλλωστε σε πολύ καλή βάση. Ορισμένοι λοιπόν κινούνται προς μια κατεύθυνση και άλλα, για παράδειγμα τα εθνικά κοινοβούλια, κινούνται προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό βέβαια είναι αναπόφευκτο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει κανείς να εγκύπτει νομοθετήματα με πάρα πολύ προσοχή και αυστηρότητα πνεύματος. Εγώ θεωρώ πάντως ότι είναι καθήκον του ευρωπαϊκού επίπεδου να συνδράμει τα εθνικά κοινοβούλια, να εξετάζουν τα θέματα εφαρμογής της επικουρικότητας, γιατί δεν έχουν τον χρόνο ούτε τους πόρους τουλάχιστον οι μικρότερες χώρες, για να μπορέσουν να ε, προβάλλουν αυτές τις ενστάσεις επικουρικότητα. Ο κύριος Ντάθ. President, um, ε, national parliaments are ε, not part of the legislative processes of the EU. Τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι τμήμα της νομοθετικής διαδικασίας της Ένωσης έχουν δικαίωμα προνομοθετικού ελέγχου μόνον με βάση την επικουρικότητα. Και τότε εκείνα αποφασίζουν πώς ακριβώς θέλουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβοηθά την τεχνική εργασία των εθνικών τιούτων, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τις χωριστές, τις διαφορετικές εντολές που έχουν τα δύο είδη κοινοβουλίων. Μερικοί ομιλητές, νομίζω, συγχαίουν αυτήν, αυτόν τον διαχωρισμό όταν μιλάνε για την εφαρμογή του, της αρχής της επικουρικότητας στην πράξη. Συμφωνώ βέβαια απολύτως με τον κύριο Ρενγκάο ότι την, σε επικρίσεις μας πρέπει να τις βασίζουμε στη συνθήκη της Λισαβόνης και όχι του Αμστελοδάμου. Αλλά διαφωνώ ότι είναι κατάλληλη εποχή τώρα για να ξαναδούμε είτε τον ορισμό της επικουρικότητας στη συνθήκη είτε τους πρακτικούς διακανονισμούς που καθόρισαν τα Εθνικά Κοινοβούλια για την εφαρμογή της. Είναι πολύ νωρίς. για να αποφανθούμε τελειωτικά για αυτό το θέμα. Χρειάζεται νομίζω, το σημαντικότερο είναι να δούμε πώς ακριβώς η Κομισιόν ανταποκρίνεται σε αυτή την πρώτη χρήση κίτρινης κάρτας. για τον λεγόμενο νόμο Μόντι 2 για την απασχόληση. Είναι λεπτό θέμα βέβαια γιατί διαχωρίζει τα κόμματα σε δεξιά και αριστερά. Και δεν είναι απλώς θέμα που διαχωρίζει κράτη μεταξύ τους. Αν δούμε τις νομοδοτήσεις που δίνουν τα εθνικά κοινοβούλια βλέπουμε ότι είναι πολύ διαφορετικής ποιότητας μεταξύ τους. Μερικές είναι καλά δομημένες και ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουμε θεσπίσει, άλλες όμως όχι. Και απλώς εκφράζουν η πολιτική τους δυσφορία ή διαφωνία ως την πολιτική της Κομισιόν. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον πώς ακριβώς θα απαντήσει η Κομισιόν στη χρήση αυτή της κίτρινης κάρτας. Την γνωμοδότησή μας νομίζω δεν πρέπει μόνο να επικρίνουμε τα εθνικά κοινοβούλια για τον μη σταθερό τρόπο με τον οποίο αντιδρούν, αλλά και την Κομισιόν που πολλές φορές πέφτει κάτω από τα νενομισμένα κριτήρια σαφήνειας, πληρότητας ή περιεκτικής εξήγησης στα μνημόνια της όταν θέλει να δικαιολογήσει τις πρωτοβουλίες της στο θέμα της επικουρικότητας. Και αυτής και της Κομισιόν δηλαδή οι γενικές διευθύνσεις ε, είναι διαφορετικής ποιότητας στις απαντήσεις τους. Νομίζω ότι το σύνολο των Επιτρόπων και ο Πρόεδρος πρέπει να δουν αυτό το θέμα για να αντιδρούν όλοι με την ίδια ποιότητα. Έχουμε λοιπόν ακόμη δουλειά με τη γνωμοδότηση αυτή. Και ίσως ο συντάκτης να πρέπει να μας εξηγήσει τι γίνεται και στη νομική επιτροπή. Πού έχει φτάσει η συγγραφή της έκθεσής τους. Ναι, κοιτάξτε στο έγγραφο της Κομισιόν για την Επιπορικότητα και την Αναλογικότητα στη σελίδα 2 λέει ότι στο μέταλ νομοθετικό επίπεδο μπορεί να επικριθεί η νομιμότητα αλλά ποτέ το δικαστήριο δεν έχει ακυρώσει καμία απόφαση με βάση την επικουρικότητα. Αυτό είναι γιατί έχουν γίνει λίγες προσφυγές ή γιατί έχει το δικαίωμα το δικαστήριο να μην το πράξει, να μην ακυρώσει. Α, δεν έχουν καταφύγει, δεν έχουν προσφύγει, μάλιστα. Α, τότε καλά. Πριν δώσω το λόγο να απαντήσει η κυρία Ρέγνερ, ο συνάδελφος Ραντζερ, θέλει να ρωτήσει κάτι τον Μπρόγκς. Θα είμαι συντομότατος. Αν μου το επιτρέπετε και αν δεν το θεωρείτε αλαζονικό, ο συνάδελφος Άγνιου πρέπει να γνωρίζει ότι επικουρικότητα είναι λατινική λέξη και προέρχεται από τη στρατηγική του Ρωμαϊκού στρατού. Δεν είναι αγγλική λέξη. Και αν μου το επιτρέπει επίσης, το όνομά σας Άγνιου έχει λατινικές ρίζες. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικοί το προφέρουν Άνιου και όχι Άγνιου. Μακρινές αλλά λατινικές ρίζες. Πρέπει λοιπόν να δεχτείτε ότι και στα αγγλικά υπάρχουν λατινικές ρίζες. Α, οι πολιτιστικές ανταλλαγές ιδίως βορρά νότου είναι πάντα κάτι που... Ε, συνάδελφε Άγνιου, Έγνιου, το λέω καλά, του δίνω, το λόγο, βεβαίως, βεβαίως. Σχεδόν όλες οι αγγλικές λέξεις προέρχονται από άλλες γλώσσες, γιατί μας έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι τόσο πολλές φορές. Το όνομά μου, περίμενε, το όνομά μου είναι μάλλον γαλλικό, από το αρνί. Και αφού είμαι γεωργός δικαιολογείται. Μα το είπα λατινικά, γαλλικά. Αλλά η λέξη επικουρικότητα δεν ακούγεται εύκολα από αγγλικά αυτιά. Το είπα και πριν. Κι όμως είναι κάτι τόσο ουσιώδες για τη διακυβέρνησή μας. Αυτό προσπαθούσα να σας πω πριν. Ωραία. Συζητήσαμε και περί ετοιμολογίας των, λέξεων, κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλους για τις παρεμβάσεις σας που βρίσκω ότι είναι πολύτιμες διότι έχετε προβεί σε πολλές συμπληρώσεις του έργου μου και χαίρομαι πολύ για την υπεραιτέρω συνεργασία. Κάτι που είναι σημαντικό για μένα και το λέω τώρα αρκετά έτσι ελαφρά ας πούμε είναι να ρέει η νομοθεσία και η επικοινωνία με τα εθνικά κοινοβούλια επίση γνωρίζοντα βέβαια ποιο ρόλο είναι ο δικό μα και ποιο είναι ο δικό του. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα την άποψη, με την άποψη μάλλον, ότι η αρχή τη επικουρικότητα είναι ουδέτερη. Δηλαδή ότι αποσκοπεί σε μια διάκριση. Για ποια πράγματα είμαστε αρμόδιοι εμεί, για ποια πράγματα είναι αρμόδιε οι εθνικέ βουλέ. Και ε, ίσω σε ορισμένε περιπτώσει είναι περισσότερα καθήκοντα, σε άλλε λιγότερα. Για μένα είναι σημαντικό στην πράξη να είμαστε ρεαλιστές. Και γι' αυτό έκανα την παραπομπή στην ε, συνθήκη του Άμστερνταμ που δεν είναι βέβαια ευανάγνωστη αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι το πρακτικό. Να εξηγήσουμε δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές οι guidelines που δεν επαναλαμβάνονται στην συνθήκη της Λισαβόνας. Βέβαια είμαι ανοιχτή σε κάθε παραπέρα συζήτηση. Η ιδέα πρόταση της κυρίας Στάιν μου, βρίσκει, φαίνεται πολύ ε, να γίνει μια ανάλυση δηλαδή και μια γνωμοδότηση και για να περιλάβει και το σύστημα IPEX που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό διότι είναι ένα πράγμα ρεαλιστικό. Και επίσης για τις μελέτες αντικτύπου, impact assessments. Αυτά και η μορφή περί επικουρικότητας είναι σαν να συγκρίνει κανείς μήλα με αχλάδια. Δεν γίνεται. Ακριβώς λέει γι' αυτό, τόνισα εγώ, επειδή η ανάλυση μου λέγεται καλύτερη νομοθεσία, better lawmaking. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεχωρίζουμε τα πράγματα και να επισημαίνουμε ότι διακρίνονται αυτό μπορεί να διευκολύνει για μια παραπέρα διευκρίνηση, όχι όμως να οδηγήσει σε συγχύσεις. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον σε συζήτηση και όλες οι παρεμβάσεις σας και επαναλαμβάνω ότι αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συνεργασία μαζί σας για να καταλήξουμε με συμπερίληψη των προτάσεών σας σε μια στέρεα θεμελιωμένη ονομοδότηση. Ο μου για την νομική επιτροπή. Ναι, ναι. Ε, ε, λυσμόνισα να σας απαντήσω. Θα ρωτήσω όμως, θα ρωτήσω. Αύριο έχουμε νομική επιτροπή. Δεν ξέρω τώρα από στήθους αν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Όμως θα σας διαβιβάσω αμέσως τις σχετικές πληροφορίες. Τα συζητούμε, αλλά δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συζήτηση αυτή. 19 Ιουνίου να ψηφίσουμε αν η νομική επιτροπή ολοκλήρωσε. Λοιπόν, εάν θέλετε να εξετάσουμε ένα θέμα το οποίο θα εξετάσαμε αύριο το πρωί, έκθεση Τρατσκόφσκι σχετικά με το θέμα της, ε, του περιεχομένου των εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε σήμερα. Υπάρχει και το σχετικό έγγραφο στο ντοσιέ. Εάν συμφωνείτε, δεν βλέπω κανένα να έχει αντίρρηση, να εξετάσουμε το την έκθεση Τσα, Τσαρσκόφσκι και παρακαλώ τον κύριο Τσαρσκόφσκι να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα που έχουμε. με αυτή τη διαδικασία. Ήταν από τις πρώτες που είχαν εφευρεθεί το 80 από την ενιαία πράξη. Αλλά από τότε άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Τώρα είναι σχεδόν άχρηστη. Η αρχική ιδέα ήταν το κοινοβούλιο να μπορεί μόνο να πει ναι ή όχι. Όταν επρόκειτο για συμφωνίες σύνδεσης ή ένταξη ή ακόμη και για μερικές εμπορικές συμφωνίες ήταν βέβαια πολύ δύσκολο να πει κανεί ναι, απλώς ναι ή όχι. Το είδαμε και με τα πρωτόκολλα όπου μπλοκάραμε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Σήμερα όμως το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια και έλλειψη συνέπειας και πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να υποφανθούμε με άλλο τρόπο, όχι ναι ή όχι. Θα έπρεπε να μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω και να εξηγούμε τη θέση μας αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα όπως πρέπει. Τώρα αν τα δούμε όλα ένα προς ένα θα χρειαστεί πολύς χρόνος, αλλά το πρώτο πρόβλημα όπου υπάρχει ασάφεια στον κανονισμό είναι το κατά πόσον η απόρριψη μιας πρότασης σημαίνει την έγκριση της αντίθετης απόφασης. Σε πολλές περιπτώσεις έτσι μας λένε ότι αν απορρίψουμε μια πρόταση τότε έχουμε de facto εγκρίνει το αντίθετο αυτόματα. Αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα διαφοροποίησης. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή δεν παίρνουμε την αλφα απόφαση ή καθυστερούμε την αλφα απόφαση για τους εξής λόγους. Δεύτερο ερώτημα και εδώ πάλι προσπαθώ να απλοποιήσω είναι το θέμα των τροπολογιών. Η διαδικασία consent, ε, της ε, έγκρισης δηλαδή, δεν προέβλεπε ούτε τροπολογίες. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα στο ίδιο το κείμενο. Αλλά το θέμα είναι μήπως δεν θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Η κάθε επιτροπή αλλιώς το βλέπει βέβαια και άλλη εναλλακτική λύση προτείνει. Παράδειγμα, σε ορισμένες επιτροπές προσθέτουν ένα ψήφισμα. Βέβαια το ψήφισμα μπορεί κανείς να το τροπολογήσει όπως θέλει. Στην ΕΠΕΞ και στην ίντε το κάνουν αυτό. άλλη ιδέα να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του προημίου και αυτό το κάνουν διάφορες επιτροπές και σε άλλες είναι πολύ αυστηρότεροι οι συνάδελφοι και δεν επιτρέπουν καμία τροποποίηση κανενός τύπου. Υπάρχει και ένα πιο πολύπλοκο ακόμη θέμα γιατί ο κανονισμός δεν διαφοροποιεί απόλυτα τη φάση της Επιτροπής με τη φάση της Ολομέλειας. Κατ' εμέ χρειάζεται καταρχήν σαφήνεια περισσότερη, γιατί είναι προφανές ότι οι διαφορετικές επιτροπές βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά και λύνουν το πρόβλημα διαφορετικά. Και άρα δεν γνωρίζουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βάλουμε τους λόγους για τους οποίους λέμε ναι ή όχι. Καταρχήν πρέπει να είναι σαφές αν η απόρριψή μας σημαίνει το αντίθετο ή απλώς λέμε ότι δεν παίρνουμε την απόφαση ή θέλουμε παράταση και αναβολή. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ενδυνάμωνε τη θέση μας και επίσης θα συμφωνούσε και με την εποχή μας, διότι η λογική του 80 ήταν να μην ε, μπερδεύεται το κοινοβούλιο σε όλα τα νομοθετικά, ενώ σήμερα μπορούμε, έχουμε περισσότερες δικαιοδοσίες και δεν ισχύει πια αυτό. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να πούμε τους λόγους μας και τώρα για τις τροπολογίες εδώ νομίζω πρέπει να δούμε τι θέλουμε. Αν συμφωνούμε ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε τη θέση μας και να πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί παίρνουμε ή δεν παίρνουμε μια απόφαση, τότε πρέπει να υπάρχει μια ενιαία διαδικασία όπου να λέμε ότι επιτρέπονται τροπολογίες ας πούμε στο προήμιο ή στα ψηφίσματα που συνοδεύουν το κείμενο ή και το σημαντικότερο το άρθρο 81 να ερμηνεύεται ομοιόμορφα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Παράδειγμα στα συνοδευτικά ψηφίσματα για ορισμένους αν υπάρχει συνοδευτικό ψήφισμα και εκεί πούμε τους λόγους μας το βρίσκουν πολύ αδύνατο. Για άλλους αρκεί. Για αυτούς που το βρίσκουν ανεπαρκές θα προτιμούσαν να τροπολογήσουν το προήμιο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε. Εγώ σας συστήνω πρώτα απ' όλα να καταργηθεί αυτή η αυτόματη διαδικασία και να υπάρχουν οι τρεις εναλλακτικέ που ανέφερα. Και έπειτα να επιτρέψουμε την κατάθεση τροπολογιών που να αποσαφηνίζουν τη θέση μας. Όχι στο ίδιο το κείμενο βέβαια, αυτό απαγορεύεται, αλλά στα συνοδευτικά. Προήμιο ή συνοδευτικό ψήφισμα που να μας επιτρέπουν να αναφέρουμε τους λόγους μας. Γιατί αν απλώς απορρίπτουμε κάτι και δεν λέμε γιατί, τότε μπορεί να υπάρξει παρερμηνία και παρεξήγηση. Υπάρχουν σημαντικές πράξεις, ιδίως οι εμπορικές συμφωνίες, στις οποίες η σαφής δήλωση και έκφραση της θέσης μας είναι τελείως απαραίτητη. Πάνω απ' όλα λοιπόν σαφήνεια, συνέπεια και σας προτείνω να σκεφτούμε την περίπτωση να έχουμε τη δυνατότητα εξηγήσεων των λόγων των πράξεών μας. Ευχαριστούμε. Τώρα ο Νταφ. Πρόεδρε. σκέφτομαι μήπως δεν υπερβάλλουμε τα πράγματα εδώ. Συμφωνώ ότι θα ήταν σημαντικό να υπάρχει μια συνεπής μέθοδος για όλες τις επιτροπές που βλέπουν τα πράγματα κάθε μία διαφορετικά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι μπορούμε και τι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε. Αλλά για την ίδια την απόφαση ως προς το κατά πόσον δεχόμαστε ή όχι μία πράξη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών ή με κάποια άλλη ενισχυμένη πλειοψηφία. Είναι φανερό ότι αν αποτύχουμε στην Ολομέλεια τότε δεν υπάρχει καμία συνένεση, δεν δίνουμε συνένεση και η απλή πλειοψηφία όχι η απόλυτη δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι μία κάποιου είδους συνένεση η διαφοροποίηση. Είναι απλώς μια αρνητική απόφαση. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι σε μερικές συμφωνίες ιδίως διεθνείς συνθήκες ή μνημόνια που να εξηγούν τη θέση του Κοινοβουλίου. Και τα κράτη-μέλη το κάνουν και αναγκάζεται όλο και περισσότερο και η Κομισιόν να το κάνει. Πρέπει λοιπόν να μπορεί το Κοινοβούλιο και εκείνο να το κάνει χρειάζεται κάποιος κανονισμός εδώ, κάποιος κανόνας, με βάση τον οποίο να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σημαντικά ερωτήματα αυτά που έθεσε ο εισηγητής και του εύχομαι καλή τύχη να βρει και απαντήσεις. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, Ταρκόφσκι, όχι. Κανένας άλλος δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Αναθέτουμε λοιπόν την εμβάθυνση του θέματος στον Ταρκόφσκι. Τελειώνουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής και θα αρχίσουμε αύριο το πρωί με την έκθεση Γκουαλτιέρη Ταρκόφσκι για την governance. Τώρα συντονιστές που θα είναι ιδιαίτερα σύντομοι. Ο συνάδελφος Γουαλτιέρη απουσιάζει και με παρακάλεσε να αναβάλω τη συνεδρίαση. Θα έλεγα λοιπόν να συζητήσουμε μόνο τα σημεία εκείνα τα οποία δεν μπορούν να αναβληθούν και είναι απλούστατα. Πέντε λεπτά λοιπόν διάλειμμα.